αρμόδιες ε, ελληνικές αρχές μου, έκαναν, μου υπέβαλαν έτοιμα άρσης ε, της ασυλίας του κυρίου Θεοδόρου Ζαγοράκη. Λοιπόν, Άλλη μια φορά η αγγλική καμπίνα. Εντάξει, λειτουργεί. Η αγγλική καμπίνα. Εντάξει, όλοι έχετε διερμηνία τώρα. Κύριε Κόμπενικ, δεν κατάλαβα τι θέλετε. Ωραία. Κύριε Κόμπερν, η έκφραση «ο πρόεδρός μου» είναι πολύ καλή. Και το μέλος μου. Okay. Ωραία. Λοιπόν, οι αρμόδιες ε, ελληνικέ αρχές, μου απέστειλαν έτοιμα για την άρση της ασυλία του κυρίου Θεόδωρου Ζαχωράκη. Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές μου έστειλαν ένα αίτημα άρση της ασυλία του κυρίου Γιάννου Σκόρβιν Μίκε. Με βάση το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού οι αιτήσει αυτές θα αποσταλούν στην ε, Επιτροπή Νομικών